Uh, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την έγκριση της διάταξης δύο παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν, ε, θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, σειρά της ημερήσιας διάταξης. Αύριο θα συναντήσουμε τον Επίτροπο Ντεκούκτ και για το θέμα των διαπραγματεύσεων, της έναρξης διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Θεωρήσαμε ότι ήταν προτεραιότητα να τον ακούσουμε καθώς ήθελε να έρθει να παρευρεθεί εδώ και είχε χρόνο, άλλαξα την ημερήσια διάταξη. Θα έρθει αύριο στις 9. Σας ε, παρακαλώ να είστε κι εσείς εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση. αναφερθεί αρχικά στην ε, τελική έκθεση που αφορά την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και την ανακοίνωση του κυρίου Ομπάμα και τον ε, ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership, θα ονομαστεί αυτή η εταιρική σχέση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να μιλάμε για εμπόριο, για επενδύσεις, είναι πολύ καλό το όνομα. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα έχουμε γενική απεργία στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε τι θα κάνετε με τις μετακινήσεις σας αν είστε μακριά από το Κοινοβούλιο. Λόγω της γενικής απεργίας. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Σημείο 2. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2013. Ο συνήθως εγκρίνονται. εκτός αν κατατεθούν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίας αυτής. Σημείο 3. Ανακοινώσεις. Έχουμε αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου, είμαστε ανοιχτό κοινοβούλιο, απευθυνόμαστε στον κόσμο, έχετε στους φακέλους σας ε, και έναν ε, κατάλογο αλληλογραφία. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Λουκρέσια του Ίστα δεξιά μου στη γραμματεία θα αντικαταστήσει τον Ερικέ Γεμινέν, ε, την Άννα Ερικέ Γεμινέν που έχει πάρει άδεια μητρότητας, προέρχεται από τη ΓΑΜΑ εμπορίου. Έτσι λοιπόν, ε, ας εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις της ε, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εμπορίου. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 4. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπουν του πίνακε Δημοκρατία Βουλγαρία και τη Ρουμανίας στο πλαίσιο προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω γνωρίζετε, όταν μια χώρα μπαίνει στην Τελωνιακή Ένωση, μπορεί να υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των δασμών με τις τρίτες χώρες γιατί μπορεί νωρίτερα να υπήρχαν χαμηλότεροι δασμοί σε σχέση με αυτούς της Ένωσης. Αυτό ισχύει για την περίπτωση Βουλγαρίας και Ρουμανίας εναντί της Κίνας. Ο κύριος Σόλτς είναι ο εισηγητής. Εδώ θα εξετάσουμε το σχέδιο σύστασης ε, για να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι η πρόταση. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω την ευκαιρία να μιλήσω γερμανικά και θα το κάνω. Δεν θα μακρηγορήσω. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω στην ε, γνωμοδότησή μου. Την έχουμε ήδη εξετάσει τον Ιανουάριο Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε το σχέδιο έκθεσης. Να τονίσω άλλη μια φορά ότι σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ, ε, για το σκοπό της, Ευρωπα... της Τελωνιακής Ένωσης. Ο σκοπός λοιπόν είναι να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές και να μην τους επιβάλλει φραγμούς. Και τώρα με αυτή τη Συμφωνία Αντισταθμιστικής Προσαρμογής έχουμε την ε, δυνατότητα να προσαρμόσουμε λοιπόν τις, τους ε, δασμούς των δύο αυτών χωρών με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ επικροτώ τη συμφωνία προσωπικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να την εγκρίνει Υπάρχει μια γνωμοδότηση, ένα σχέδιο έκθεσης από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο είναι προβλέπεται να εξεταστεί και να ψηφιστεί τον Μάρτιο. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι μέχρι τώρα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα υπογραφούν επίσημα αυτά τα σύμφωνα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι πιστεύω πως θα έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι εμείς να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας και να περιμένουμε μέχρι την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αυτά προς το παρόν. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά όλους και τη Γραμματεία για την υποστήριξη της αυτό το σχέδιο έκθεσης και ε, θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σας ή ενδεχόμενα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή επί... πρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια των σκιώδων εισηγητών. Ευχαριστώ. Σίγουρα αυτή η συμφωνία δεν ε, δόθηκε επίσημα στο Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε λοιπόν να την ψηφίσουμε ακόμα. Δεν έχει υπογραφεί, όπως είπατε, και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές, το Συμβούλιο θα μας στείλει τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα στείλει τη συμφωνία, και θα την ψηφίσουμε μετά την υπογραφή. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων πρώτα και σε αυτό το στάδιο να αναμένουμε εξελινήξεις. Κύριε Λάνια, έχετε σχόλια ή κάποια άλλα μέλη ενδεχομένως έχουν σχόλια. Ναι, απλώ να σας πω ότι υποστηρίζουμε απόλυτα αυτή την ε, πολύ σημαντική αλλά και τεχνικού χαρακτήρα έκθεση. Ε, Ο κύριος Ζερόμου πέρα από την Κομισιόν. Ναι, Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα στις ε, σαφέστατες εξηγήσεις του εισηγητή. Απλώς αναφέρω ότι η γραμματεία του Συμβουλίου είναι σε στενή επαφή με τους Κινέζους. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία για την υπογραφή αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά είμαστε πρόθυμοι να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Ελπίζουμε ότι θα λάβει χώρα τις επόμενες μέρες εβδομάδες. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Να προχωρήσουμε από τον εισηγητή τελικές παρατηρήσεις. Όχι, περνάμε στο σημείο 5. εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Εδώ έχουμε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών, που είναι υπεύθυνη επιτροπή και ο κύριο Στάρντι είναι ο συντάκτης της γνωμοδότησης, ήδη έχετε στο φακελό σας το σχέδιο του κειμένου. Εδώ θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στάρντι για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση σε κάτι που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι ο Κάρελ Ντεγκούχτ θα έρθει να συμφωνήσει την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμπορίου. Είμαστε νέα άτομα εδώ. Την προηγούμενη φορά στου συντονιστέ συζητήσαμε την επίσκεψη στι ΗΠΑ και θα επιτραπεί στην Επιτροπή μα να έχει μόνο πέντε μέλη στην αντιπροσωπεία. Είναι ε, αποστολή εμπορίου. Καταλαβαίνω ότι ε, έχετε συγκεκριμένη στάση, αλλά θεωρώ ότι είναι πονίδιστο το γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε μόνο πέντε μέλη σε μια τόσο σημαντική αποστολή στι ΗΠΑ. Ελπίζω να πιέσουμε ε, τα μέλη για να μπορέσει να γίνει κάτι από αυτού. Ε, ευχαριστώ ε, και οι συντονιστές και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αναλάβουν τα ενία και να πιέσουν στην διάσκεψη των Προέδρων ώστε να γίνει αλλαγή. Και εγώ φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ από πλευρά μου, αλλά νομίζω ότι χωρίς τη στήριξή σας είναι ανώφελο να προσπαθήσω μόνος μου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έθιξα το θέμα αυτό και ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Καταρχά, να, σκιώσω, να ευχαριστήσω του σκιώδει συζητητέ. Κάναμε μια συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνεισφορά του, κυρίω από τον σοσιαλιστή συνάδελφο. Θα προσπαθήσουμε να καταθέσουμε κάποιε τροπολογίε στη γνωμοδότηση για να λάβουμε υπόψη ε, τα ε, όσα προτάθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, θα καταθέσω τροπολογίε για να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η ε, αεροπλοεία στην ε, οι αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, βοηθούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Αναφερόμαστε συνεχώς σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και αερομεταφορές δραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να απογειώσουμε την οικονομία, γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις ε, να ανθίσουν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, τον ανταγωνισμό έξωθεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, και το θέμα της γλώσσας που τονίζει, συγγνώμη, να τονίσουμε κάτι το οποίο τονίζει το ρόλο της περιφερειακής αεροπορίας. Δεν το είχα αναφέρει αυτό αρχικώς στο σχέδιο ε, της πρότασής μου. Ε, κάποιοι πρότειναν να αναφέρω και το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ε, την αναστολή των διαπραγματεύσεων στον ε, Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, τον ICAO. Θα υπάρξει σχετική διατύπωση από αυτό. και έχω κάποιους δισταγμούς για τις τροπολογίες που αφορούν το, τη ρήπανση, την ηχορύπανση. Ε, δεν θα ήθελα να συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεσή μου, διότι ε, δεν ε, ε, περιλαμβάνεται κατά την άποψή μου στο πεδίο εφαρμογή τη γνωμοδότηση τη ΣΥΝΤΑ. Αυτή είναι η θέση μου βέβαια. Μπορείτε εσεί κάλλιστα να καταθέσετε τροπολογίε. Κατάθεση τροπολογιών τελική ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου. Προσβλέπω στι τροπολογίε σα. Ωραία, να δώσουμε το λόγο στου κοιόδη εισηγητέ. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο πρώτος? Η κυρία Σαρνέζ. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση. Δεν ε, έχουμε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης ε, τη σήμερον ημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως ο τομέας των αερομεταφορών είναι μια δυνατότητα ανάπτυξης. Ίσως θα έπρεπε στο σημείο 2 να ενισχύσουμε ε, το θέμα αυτό. ξέρω ότι και εσείς θεωρείτε την ευκαιρία, καλό θα ήταν να αναφέρετε. Για το σημείο 3 να πω κάποια πράγματα. Λέτε ότι θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα ευρωπαϊκά μέσα. Μήπως θα έπρεπε να αναπτύξουμε νέα μέσα ερωτηματικό είναι αυτό. Εσείς ε, θα δείτε ε, αν μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στον τομέα των αερομεταφορών. Και επίσης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στο θεμητό ανταγωνισμό, στο δίκαιο ανταγωνισμό και εγώ θεωρώ ότι είναι καλό ότι το αναφέρεται εδώ. Για το σημείο 4 νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην καταπολέμηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι περισσότερο εκτός από το να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο ε, ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τον ηγετικό ρόλο εδώ για να έχουμε ένα καλύτερο διεθνές ε, νομικό πλαίσιο στο θέμα αυτό, όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας και με τους δύο όρους, αλλά και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Για το σημείο υπαριθμών 7 γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ε, ε, τη ε, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ίσως θα έπρεπε να τις αναφέρουμε αυτές. Ε, οριστικοποιήθηκε και η συμφωνία με τη Βραζιλία και ίσως θα έπρεπε να προσθέσουμε και την Ιαπωνία, και πάλι ερώτηση είναι αυτό, εν ώψη των ε, διαπραγματεύσεων για μια συνολική συμφωνία. Μήπως θα έπρεπε ίσως και στη γνωμοδότηση να αναφέρουμε και κάτι για τις ε, ε, διασταυρούμενες επενδύσεις, δηλαδή τη δυνατότητα να ενθαρρύνουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε όθηση για διεθνείς επενδύσεις στον τομέα των αερομεταφερών. Παρακαλώ, κάποιο σκιώδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ σε ένα, στο σύνολο των σημείων, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάμε κάποιο ε, πιο μακριά σε ό,τι αφορά τον άνθρακα και την αεροπλοΐα. Προφανώς ε, ότι η υποχρέωση μείωσης ε, των εκπομπών ε, υπάρχει σε ένα τομέα που βλέπουμε ότι μεγεθύνεται έτσι λοιπόν ε, η καινοτομία εδώ στον τομέα των εκπομπών του εξή του άνθρακα είναι κάτι σημαντικό στο με της και η αγορά του άνθρακα είναι ίσως ε, ενδυνάμει μια πηγή εσόδων για τα κράτη. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια αγορά άνθρακα στα 30 δολάρια τον τόνο και τα επόμενα 7 χρόνια την επόμενη περίοδο θα φτάσουμε περίπου στα 200 ε, ε, δισεκατομμύρια δημοσίων εσόδων που θα μπορούσαμε να έχουμε και μου φαίνεται δύσκολο να ε, εξηγήσουμε στους πολίτες ε, ότι όταν γεμίζουν με βενζίνη το αυτοκίνητό τους πληρώνουν τόσους φόρους για τον άνθρακα, ενώ όταν παίρνουν το αεροπλάνο δεν πληρώνουν τίποτα, δεν πληρώνει κανεί τίποτα για τον άνθρακα και για την κυρσίνη. Και ξέρετε ότι με αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά ε, μπήκε η αεροπλοία σε ένα σύστημα ε, κατά κάποιο τρόπο φορολόγηση. Γι' αυτό και ήταν θετικέ οι εταιρείε στο να υπογράψουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρχει μια συζήτηση σήμερα σε διεθνέ επίπεδο, είναι γιατί η Ευρώπη ήθελε να έχει ηγετική θέση. Αν τώρα η Ευρώπη αρχίσει να λέει Α, όλα αυτά θα αμφισβητήσουν την ανταγωνιστικότητά μα, δεν θα υπάρχει πλέον συζήτηση και θα σταματήσουν εκεί τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τη συνάδελφο την ε, Μαριέλ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε κάπως ε, πιο ισχυροί να έχουμε πιο κάθετη άποψη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Σκιώδη εισηγητή, γιατί δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, είχε άλλες υποχρεώσεις, ήταν σε άλλη επιτροπή. Να προσθέσω όμως ότι στηρίζω έντονα τα σχόλια της κυρίας Δεσάν και του Γιάννικ για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην όλη συζήτησή μας εδώ για, τις, για ε, το εμπόριο εκπομπών. Μία ερώτηση όμως να κάνω. Ο κύριος Στέρντι μόλις ανέφερε ότι δεν θέλει να συμπεριληφθεί η μείωση των θορύβων στη γνωμοδότηση. Εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε αντίθετα να υπάρχει, διότι και αυτό είναι ζήτημα ανταγωνισμού. Δείτε τους πολίτες και το πώς εκείνοι επηρεάζονται όσοι μένουν κοντά σε αεροδρόμια από τα αεροπλάνα που απογειώνονται και προσγειώνονται. Η μείωση των θορύβων ε, λοιπόν γίνεται πρόβλημα εκεί που υπάρχουν τα αεροδρόμια όπου έχουμε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις πόλεις, στα αεροδρόμια. Είναι ζήτημα η, η χορύπανση και οι πολίτες επομένως πρέπει και εκείνοι να συμφωνήσουν για την αύξηση των, ε, του όγκου των αερομεταφορών, διότι πιστεύω πως αυτό το ζήτημα είναι διεθνές, αφορά όλους και η αύξηση των ε, αερομεταφορών επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών που ζουν σε περιοχές ε, κοντά σε αεροδρόμια και πιστεύω λοιπόν πως για αυτούς τους λόγους πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό. Ευχαριστώ. Κύριος David Μάρτιν. Ναι, θα είμαι σύντομο. Ο Ρόμπερτ είπε κάποια στην εισαγωγή του, αλλά δεν το βλέπω στην ε, γνωμοδότηση για τα περιφερειακά αεροδρόμια και πιστεύω ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι πολύ σημαντικά από εμπορικής ε, άποψης. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να βάλουμε όλες τις μεταφορές στα κομβικά αεροδρόμια, στα πολυκεντρικά, αλλά τα περιφερειακά αεροδρόμια θα έχουν, έχουν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στον τομέα αυτό και πιστεύω πως εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν, γνωρίζω, δεν ξέρω ακριβώ πώς θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε, αλλά ίσως θα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την συγκέντρωση των, ε, του όγκου κάπως. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Επιτροπή, διότι αυτή η έκθεση βασίζεται σε μια ανακοίνωσή σας κύριος Κλάους Γκάιλ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σαφέστατο και σύντομο σχέδιο έκθεσης και σας ευχαριστούμε και για την υποστήριξη για τα κυρία συμπεράσματα της Κομισιόν που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή τη. Πράγματι, η αεροπλοεία δραματίζει ένα στρατηγικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και για την ε, μεγέθυνση και για τη συνθεσιμότητα με ολόκληρο τον κόσμο και τη δημιουργία θεσμών Έχει ρόλο βασικό για το διεθνέ εμπόριο, αλλά και για τη δημιουργία επαφών μεταξύ των χωρών παγκοσμίω. Έχουμε ένα καλό ρεκόρ στην αεροπλία. Σήμερα έχουμε τρει από τι μεγαλύτερε αεροπορικέ εταιρείε στον κόσμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τρει από του μεγαλύτερου αεροπορικού κόμβου και ο κλάδο ε, υποστηρίζει πάνω από 5 εκατομμύρια θέσει εργασία ε, και συνεισφέρει πάνω από 350 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ. Πάνω από 2% δηλαδή. Επίση έχουμε ηγετική θέση στην κατασκευή αεροσκαφών και μηχανών, αλλά καμία από αυτές τις ε, ηγετικέ θέσεις ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Και σε πολλούς ε, τομείς οι θέσεις μας απειλούνται από νέες προκλήσεις στα πλαίσια ενός πιο ανταγωνιστικού κλάδου. Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση του Ευρωπαϊκού Τομέα Μεταφορών, πρέπει να κάνουμε πιο φιλόδοξη την πολιτική μας και θα πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει στρατηγική. Για πολλά χρόνια υποφέραμε από κατακαιρματισμό σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε πάρα πολλές διμερείς ε, συμφωνίες. Επομένως, είμαστε ικανοποιημένοι με τα συμπεράσματα που κατέρτισε ήδη το Συμβούλιο από την ανακοινωσή μας, ε, που καταρτίζουν έναν ε, χάρτη πορείας για, μια πιο φιλό, για ένα πιο φιλόδοξο κλάδο μεταφορών τα επόμενα έτη. Θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε καθολικές συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις ε, όμορες χώρες εντάσσοντας τις γειτονικέ χώρες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών ε, βάση υψηλών προτύπων, υψηλής προστασίας, ε, ασφάλειας και σε τομείς κοινωνικής εργασίας. Επίσης, θα επιδιώξουμε συμφωνίες με βασικούς εταίρους, όχι μόνο με τις όμορφες χώρες, αλλά και με νέες αναδυόμενες αγορές, όπως οι χώρες BRICS. Επίσης, έχουμε ήδη συνολικά καθολικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Διαπραγματευτήκαμε μια συμφωνία με τη Βραζιλία. Όμως, δυστυχώς, η Βραζιλία δύο χρόνια μετά τη μονογράφηση της συμφωνίας, επανήλθε και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση σε αρκετά σημεία, τα οποία τώρα συζητούμε στο Συμβούλιο. Γιατί αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια διευρυμένη εντολή για να συνάψουμε τη συμφωνία με την Βραζιλία, που νομίζουμε ότι είναι μια στρατηγική αγορά για τις ε, εταιρείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν λάβουμε και υπόψη ότι τα επόμενα έτη θα φιλοξενήσει η Βραζιλία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τη σημασία που προσδίδει ο συζητητής ε, στην ε, διαφύλαξη του ασφαλούς ανταγωνισμού Έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των ε, εταιρείων μεταφορίας στον περσικό κόλπο όπως η Emirates, η Qatar Airways. Είναι καλό αυτό για τις μεταφορές, ε, αλλά δεν είναι καλό απαραίτητα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Και ακόμη και οι ευρωπαϊκοί κόμβοι βλέπουν ε, να μειώνεται η κυκλοφορία σε αυτούς τους κόμβους ε, υπέρ κόμβων ε, στον κόλπο. Και ο ανταγωνισμός ε, με τις εταιρείες αερομεταφορών στην περιοχή αυτή δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερα διαφανής και έχουμε ανησυχίες για τον θεμητό ανταγωνισμό. Κάποιος βουλευτής ανέφερε μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί ένα νέο μέσο προς αυτή την κατεύθυνση και σκεφτόμαστε πράγματι όχι μόνο αναθεώρηση τον σημερινό ε, μηχανισμό εμπορικής άμυνας, αλλά και ένα πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για να διασφαλίσουμε το θεμητό ανταγωνισμό. Και αυτές τις προτάσεις θα τις παρουσιάσουμε του επόμενους μήνες. Επίσης αναφέρθηκε ότι η Κομισιόν έχει εντολή να διαπραγματευτεί με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Έχουν ε, παγώσει Αυτές οι διαπραγματεύσεις για διάφορους λόγους θα θέλαμε να ολοκληρωθούν. Επίσης έγινε αναφορά σε διασυνοριακές επενδύσεις στον τομέα της ε, αεροπλοείας, στον τομέα των ερμητοφορών. Αυτό θα το καλωσόριζε η Κομισιόν. Σήμερα ο παγκόσμιος κλάδος μεταφορών ε, τεχνικά υποδίζεται από εθνική σημαντικούς περιορισμούς ε, για τον έλεγχο των εταιριών ε, και αυτό περιορίζει την πρόσβαση των εταιριών ε, στο κεφάλαιο, στη χρηματοδότηση. Για κάποια σχόλια που έγινε σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. όπω ξέρετε, η Κομισιόν πριν κάποια χρόνια πρότεινε τη συμπερίληψη των ερμετοφορών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα ETS, γιατί ξέρετε ότι αυξάνονται οι από τον τομέα των ερμετοφορών. Αυτό έχει δημιουργήσει έντονες συζητήσεις ε, σε όλο τον κόσμο και τη αντιδράσεις από Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, ακόμη και ΙΠΑ. Αλλά η πρόσφατη πρόδρος ε, που έγινε με τις συζητήσεις στον ΙΚΑΟ για την αναζήτηση παγκοσμίων μηχανισμών με βάση της αγοράς ε, για την ε, αντιμετώπιση των ε, κλιματικών αλλαγών των, περιβαλλοντικών συνεπειών προέρχονται από το μεταφορών μας έχει ενθαρρύνει. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και τώρα η Κομισιόν έχει ενθαρρυνθεί από την πρόεδρο που έχει γίνει τελικά σε, σε παγκόσμιο επίπεδο και θα δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στην ε, συνεδρίαση του ΙΚΑΟ. Προσπαθούμε εμείς να έχουμε ηγετική θέση στη συζήτηση εκείνη, προκειμένου να πετύχουμε καλά αποτελέσματα και για την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, θα ολοκληρώσω εδώ και πάλι ευχαριστώ τον Σιγητή για μια εξαιρετική έκθεση. Ξεκάθαρα στην έκθεση αυτή ζητάτε μια πιο φιλόδοξη και συναφή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μέτρων Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες και να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση με τον εισηγητή μας, ο κύριο Στέρντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας παρακαλώ στείλτε μου τις παρατηρήσεις σας ε, είτε με, ε, σε μορφή τροπολογίας ή όπως ακριβώς επιθυμείτε. Και ο Γιάννη και ο Χέλμερ. Να πω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχω συμπεριλάβει πολλές από τις προτάσεις που κάνετε είναι διότι ήθελα η συγκεκριμένη ε, γνωμοδότηση ε, να ε, επικεντρωθεί στα θέματα εμπορίου. Συμφωνώ όμως με όλα όσα είπατε, δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση και είμαι βέβαιος ότι καταθέσετε και σχετικές τροπολογίες. David, έχεις δίκιο. Δεν ήταν στην αρχική έκθεση, θα έπρεπε να είναι. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που μου διέφυγαν μάλλον. Αλλά ανέκυψε στη συζήτηση στο Στρασβούργο και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο γίνονται οι συνεδριάσει με του κοιόδη ηγητέ για να γίνεται αυτή η πολυδοσκόπηση και να παίρνουμε ιδέε. Συμφωνώ μαζί σου, είναι ζωτική σημασία και συγγνώμη που δεν το ανέφερα, αλλά θα τροποποιηθεί και αυτό ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάπου θα το συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Ωραία, ευχαριστώ. Θα έχουμε μια εξαιρετική γνωμοδότηση λοιπόν. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου. Κάντε λοιπόν τις προτάσεις σας. Τώρα, για να περάσω στο προηγούμενο θέμα, μου ζητήθηκε να ανακοινώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση του Χέλμουντ Σόλτς για την ε, σύστασή μας για τη συμφωνία με την Κίνα, γιατί δεν θα ψηφίσουμε μεν, αλλά θα πρέπει να καταθετεθούν τροπολογίες. Προθεσμία λοιπόν κατάθεσης τροπολογίων 1η ε, Μαρτίου. Σημείο παριθμών 6. εμπόριο μεταξύ ε, κοινότητας και τρίτων χωρών για πρόδρομες ουσίες ε, φαρμάκων. Είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Η συγητής είναι ο Φρανκ Προύστ από το ΕΛΚ. Το σχέδιο έξεθεσης περιλαμβάνεται ήδη στο φάκελό σας και θα γίνει η συζήτηση επί του σχεδίου εκθέσεως. Πρόκειται για ένα ε, θέμα το οποίο θέλει να τροποποιήσει τον κανονισμό 111 του 2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών και θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τον κανονισμό και να ευθυγραμμίσουμε τον κανονισμό αυτό με τις ε, κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις βάσει των όσων ισχύουν ε, αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό. Εδώ είναι ο συγητής μας και θα του δώσουμε αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως θα διαπιστώσατε, ε, έχω τροποποιήσει λίγο την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού για το εμπόριο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Η βασική τροποποίηση που έχω κάνει είναι ότι έχω συμπεριλάβει στις ε, ε, ουσίες που περιλαμβάνονται στην κατάταξη και τα φάρμακα. Εξηγώ στην αιτιολογική μου έκθεση ότι μέχρι τούδε στην πρόταση τροποποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα φάρμακα αποκλείονται από το πεδίο διαβαθμισμένες ουσίες. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ένα φάρμακο χρησιμοποιείται όμως ε, για να ε, παρασκευάσουμε ναρκωτικές ουσίες, θα πρέπει να περάσουμε από τη διαδικασία συναπόφασης για να ε, θεωρηθεί ότι δεν πρέπει να εισάγεται η συγκεκριμένη ουσία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα καθυστερήσουμε περίπου δύο χρόνια πριν μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών και δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Προτείνω λοιπόν να συμπεριλάβουμε ε, στις διαβαθμιμένες ουσίες και φάρμακα των οποίων μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε κάποιες πρόδρομες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζεται μόνο μία κατεξουσιοδότηση πράξη για να ε, ε, μπορέσουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τις ουσίες αυτές και έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα τάση των ε, εμπόρων ναρκωτικών και ε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα φάρμακα αυτά. Ε, θα μπορέσουμε να τις περιλάβουμε λοιπόν αν μια ουσία περιλαμβάνεται στο φάρμακο και μπορούμε εύκολα να την εξάγουμε, ε, να τη βάλουμε στις διαβαθμισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η εφεδρίνη και η ψευδροεφεδρίνη. Ε, δεν θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε προβλήματα και για όσους φοβούνται ότι μπορεί να ε, δημιουργήσουμε προβλήματα στο εμπόριο των πρόδρομων ουσιών που είναι πολύ σημαντικό για κάποιες ε, τρίτες χώρες να σας πω ότι η εφεδρίνη και η ψευδοεφεδρίνη είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αλλεργιών και κρυολογημάτων επομένως είναι φάρμακα που βρίσκονται εύκολα. τα φάρμακα τα οποία περιέχουν εφεδρίνη και ψευδεφεδρίνη ε, έχουν μια πολύ ε, τυπική διαδικασία έγκρισης και ε, με βάση την αξιολόγηση επιπτώσεων το κόστος τους είναι περίπου 15 ευρώ. Ε, κανονικά θα έπρεπε σε αυτή την κατηγορία να συμπεριλάβουμε και άλλα φάρμακα από αυτά τα ήπια τα οποία σας ανέφερα. Επίσης, η δεύτερη τροποποίηση που θα ήθελα να κάνω σε αυτόν τον κανονισμό αφορά τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Θα ήθελα οι εκτελεστικές πράξεις να ακολουθούν μια διαδικασία διαβούλευσης που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία διότι η καταπολέμηση της εμπορίας των ναρκωτικών δικαιολογεί μια τέτοια στάση. Προτείνω κάποιες συγκεκριμένε ε, ε, διατάξεις για το τι γίνεται με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο 5 ετών και να μην είναι ε, επαόριστον αυτή η εξουσιοδότηση. Ελπίζω να μην σας καθυστέρησα και προσβλέπω στα σχόλιά σας. Thank you for your... Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Πραγματικά εκτενής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, εδώ μιλάμε για την αναθεώρηση ενός κανονισμού που φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις τροπολογίες, γιατί νομίζω προς την κατεύθυνση αυτή πηγαίνουν. Και ίσως αυτό που θέτει η Κομισιόν θα ε, μπορούσε ίσως να αλλάξει την κατάσταση για την κατάχρηση ουσιών ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ναρκωτικών. Όμω θέλω να ρωτήσω κάτι την Κομισιόν για να μα το διευκρινίσει, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια νομικά κενά σε ό,τι αφορά τις κοινοποίησεις παραδείγματος χάρη, αν ε, ένα προϊόν ή φάρμακο που θα μπορούσε να έχει καταχωρηθεί στις ομάδες 1, 2 ή 3 χρειάζεται άδεια εξαγωγής αλεφιδρίνη και ψευδεφιδρίνη. Δεν χρειάζονται αυτή την κοινοποίηση, ούτε οι έμποροι χρειάζονται άδεια. Θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια παράδοξη κατάσταση. Ο εισαγωγέας ε, ο οποίος ε, ενημερώνει εκούσια τις αρμόδιους φορείς ότι θα κάνει μια εξαγωγή, ε, μπορεί να κάνει αυτή την εξαγωγή ή όχι, αλλά αν την κάνει έχουμε πρόβλημα με το τελευταίο. Τι κάνουμε δηλαδή με το πακέτο που έχει παρακρατηθεί, ποιες είναι οι νομικές εγγύησεις και πώς ακριβώς τεκμηριώνεται η διακράτηση αυτού του πακέτου και τι συμβαίνει με το κόστος, με τις δαπάνες. Αυτό πάντοτε απασχόλησε ε, και την Κομισιόν αλλά και εμάς. Γιατί δημιουργούνται έξοδα για τα κράτη μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν κάποια νομικά κενά που θα έπρεπε να τα ξεκαθαρίσουμε για να μην έχουμε ανασφάλεια δικαίου. Νομίζω ότι η ταχύτητα που θέλει να δοθεί στον κανονισμό είναι κάπως αμφίσιμη αν ε, δεν προσδιορίσουμε τα θέματα αυτά συγκεκριμένα. Να δούμε δηλαδή τι θα κάνουμε συγκεκριμένα στην πράξη. Γι' αυτό απευθύνομαι στην Κομισιόν. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος κοιόδης. Η Φραντσίσκα Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως εδώ πρέπει να δούμε επίσης και το όλο ζήτημα του τι προτείνει η Επιτροπή, να το δούμε αναλογικά. Διότι αν όλες αυτές οι εταιρείε πρέπει να καταχωρηθούν, πρέπει να αναρωτηθούμε και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις ίδιες τις εταιρείε και τους χρήστες των φαρμάκων τα οποία περιέχουν τις ουσίες αυτές. Δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά και στους καταναλωτές και στην τιμή των φαρμάκων και στις ε, ενδεχόμενες καθυστερήσεις της ε, παραδώσει των φαρμάκων στην αγορά. Εμείς δεν συμφωνούμε με την διεύρυνση του ε, ελέγχου, όπως προτείνει ο εισηγητής. Αντίθετα, πιστεύουμε πως αυτό δεν θα ήταν καλό. Δεν θα ήταν καλό να διευρυνθεί ο έλεγχος και να προσθεθούν νέες απαιτήσεις πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τη λιγότερη δυνατή, τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες. Συνοψίζοντας να πω ότι χάρηκα πολύ που άκουσα τις απόψεις της Επιτροπής και θα υποβάλουμε τις δικές μας τροπολογίες. Μάλιστα, με εκπλήσει που η πράσινη είναι αντίθετη σε διεύρυνση του κανονισμού. Πολ Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όσον αφορά το πώς επηρεάζει τους καταναλωτές, ε, να σας πω ότι έχουμε να κάνουμε με τις μεθαμφεταμίνες και την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Υπάρχει αύξηση της χρήσης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω πως ε, η απαγόρευση από μόνη της δεν κατάφερε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και να σας πω ότι όλα αυτά επίσης είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις επιπτώσεις της κρίσης, με την καταστροφή των κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών. Να δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Ελλάδα όπου υπάρχει ύφεση και λιτότητα. Δείτε πώς συσχετίζονται οι συνέπειες της κρίσης με την σημαντική αύξηση των ε, εξαρτημένων τοξικομανών, με την σημαντική αύξηση των ε, φορέων του HIV και με την, ε, με την αλλαγή των ναρκωτικών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, που προχωρούν, απολάζουν από ηρωίνη σε κρυσταλλική μεταθαμφεταμίνη λόγω της τιμής. Δείτε τα λοιπόν αυτά και Πιστεύω πως έτσι θα δείτε πως πρέπει να αποτρέψουμε την ε, μεταστροφή των παραγωγών στην παραγωγή ε, κρυσταλλικής μεταφεταμίνης. Η προσέγγιση του εισηγητή, εκείνη της διεύρυνσης ε, δηλαδή του να γίνει πιο δύσκολη πρόσβαση στις πρόδρομες ουσίες, έχει τη λογική της. Είναι λογική με αυτό, διότι ασχολείται με το πώς ε, παρασκευάζονται τα ναρκωτικά. Αυτό αλλάζει συνέχεια. Και μπορεί σήμερα να είναι η εφεδρίνη και η ψευδοεφεδρίνη, αλλά αύριο να είναι κάποια άλλη πρόδρομη ουσία. Και αναφέρονται μελέτες όπου διαπιστώνεται αυτή η αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, χρειαζόμαστε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες, ε, αλλά θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν στηρίζει αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Αν όχι, τότε να ακούσουμε την Επιτροπή. Όχι μόνο επειδή εκείνοι συνέταξαν την πρωτοβουλία, αλλά και επειδή διατυπώθηκαν πάρα πολλέ ερωτήσει προ αυτού. Η Καρολίν Έντερη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια και στην έκθεση, αλλά και να απαντήσω στις ερωτήσεις που θέσατε. Πιστεύω ότι από τη συζήτηση φάνηκε πως πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισορροπία της ε, διευκόλυνσης δηλαδή του μαλλίου εμπορίου και την αποτροπή της διοχέτευσης των πρόδρομων ουσιών για παράνομες ενέργειες. Αυτό είναι κάπως δύσκολο το τελευταίο. Καταρχάς να πω ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού σε όλα τα φάρμακα δεν ήταν αυτό που εμείς επιθυμήσαμε στην αρχή, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχει ήδη μια οδηγία η οποία ρυθμίζει την παραγωγή και, την, ε, το εμπόριο των φαρμάκων. Και η οδηγία αυτή είναι αρκετά περιοριστική, διότι όλη η παραγωγή πρέπει να είναι καταχωρημένη στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα στους παραγωγούς και στους εμπόρους οι οποίοι ήδη ελέγχονται αυστηρά από αυτό το πλαίσιο. Αυτό που θέλουμε είναι να περιορίσουμε την ε, παράνομη παραγωγή ναρκωτικών με τον κανονισμό αυτό και βλέπω ότι και ο εισηγητής έχει επίγνωση της ανάγκης να μην επιβληθεί περαιτέρω φόρτος στους ε, παραγωγούς. Θα βάλουμε λοιπόν στο παράρτημα μία αναφορά στα νέα φάρμακα. Πιστεύω πως ε, αυτή είναι μία λογική προσέγγιση. Ίσως το μόνο πρόβλημα που εντοπίζω με αυτήν την ε, πρόταση είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στον ορισμό των ουσιών αυτών που καλύπτουν τα φάρμακα και τα μέτρα που προτείνονται για τον έλεγχο των φαρμακών αυτών. Στο άρθρο 11 διαβάζουμε ότι υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για τα προϊόντα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στην διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τα προϊόντα της κατηγορίας 4. Και αυτό δεν διαφαίνεται από το κείμενο. Τώρα, Ε, όσον αφορά την ερώτηση για τα κενά που ανέφερε η κυρία Μπαριά, τα κενά στο σύστημα. Ε, στην εκτίμηση αντικτύπου υπάρχουν πολλές επιλογές. Μία από αυτές μας επιτρέπει έναν πλήρη και σωστό έλεγχο των εξαγωγών των προϊόντων αυτών για να αποφύγουμε λοιπόν τη, την παράνομη χρήση τους. Γιατί λοιπόν να επιβαρύνουμε περισσότερο το διοικητικό φορτίο. Όπως είπαμε και πριν, οι παρασκευαστές φαρμάκων είναι ήδη καταχωρημένοι σε Μητρώα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επιβαρύνουμε ούτε εκείνους ούτε τις αρχές περισσότερο. η εξαγωγή φαρμάκων που περιέχουν εφεδρίνη και ψευδοεφεδρίνη γνωρίζουν ότι πρέπει να, έχουν μια πρέπει να στείλουν μια ειδοποίηση για τις ουσίες αυτές προτού εξάγουν τα προϊόντα τους. Πρώτα λοιπόν ε, αποστέλλεται αυτή η ειδοποίηση πριν την εξαγωγή και μετά δίδεται η άδεια τους δίδεται η άδεια και με την άδεια αυτή πηγαίνουν στο τελωνίο και εκτελωνίζονται τα προϊόντα τους. Φυσικά βέβαια θα πρέπει να ενημερώσουμε και τους ε, παρασκευαστές αλλά και τις αρμόδιες αρχές και είναι πολύ σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να συνεργαστούν με τα τελωνία. Δεν με ανησυχεί λοιπόν ενδεχόμενος επιπλέον φόρτος στη δουλειά τους. Επίσης ε, αναφέρατε την νευροεφεδρίνη. Γνωρίζουμε ότι τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία αυτή στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν και για παράνομη κατασκευή, παραγωγή ναρκωτικών, αλλά αυτό το έχουμε συμπεριλάβει και στον κανονισμό. Τώρα, μερικά επιπλέον σχόλια για το σχέδιο του κανονισμού αφορά την, ε, την, ε, τις πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 38, οι πράξεις αυτές έχουν περιοριστεί στην δυνατότητα μόνο να συμπεριληφθούν οι ουσίες αυτές στο παράρτημα, αλλά να μην αποσύρουμε να μην αφαιρέσουμε τις ουσίες αυτές λοιπόν από το παράρτημα, όμως ενδεχομένως θα πρέπει να αφαιρέσουμε κάποιες ουσίες οι οποίες δεν θα χρειαστεί να ε, υποβληθούν σε έλεγχο. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι αναγκαίο να μπούμε σε άλλη μια διαδικασία συναπόφασης για να αφαιρέσουμε τις ορισμένες ουσίες από τον κατάλογο. Τέλος, όσον αφορά τον χρονικό περιορισμό, τα πέντε χρόνια δηλαδή για τις, για τις ε, εξουσιοδότηση, για μας αυτό δεν είναι αρκετό, διότι χρειάζεται να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο να αντιδράσουμε στις ε, τάσεις της εμπορίας ε, ναρκωτικών και πιστεύουμε ότι το χρονικό αυτό διάστημα ενδεχομένως μας ε, επηρεάσει στην ικανότητα αντίδρασης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναθεωρήσετε τα 5-7 χρόνια και να σκεφτείτε να το αλλάξετε σε αόριστο χρόνο. Επίσης, αυτό ισχύει και για τα τελωνία. Αυτά προς το παρόν και περιμένουμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις μας το συντονομότερο. Ο εισηγητής. Uh, any to Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον εισηγητή, παρακαλώ. Ναι, μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Και αυτή η δήλωση από την πλευρά των εμπορευμένων θα ήταν ε, εθελοντική. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Όχι για να υπάρχει έγκριση της εξαγωγής πρέπει να υπάρχει πρώτα η κοινοποίηση της προεξαγωγής προς τη χώρα προορισμού. Μέσα σε 50 μέρες μπορεί να απαντήσει η χώρα και αν απαντήσει θετικά τότε θεωρείται νόμιμη η αποστολή. Αν δεν έχουν απαντήσει μπορούμε να προχωρήσουμε με την εξαγωγή. Είναι υποχρεωτική η διαδικασία λοιπόν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Ισηγητά, υπήρχαν πολλέ αντιδράσει στην εκθεσή σα. Έχετε σχόλια. Να πω δύο λόγια για την ασφαλεία δικαίου. Άκουσα τα όσα είπαν εσκιώδεις συζήτητες ε, και η Κομισιόν. Θα έχουμε το χρόνο να ξανασυναντηθούμε για να δούμε Πώ θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον κύριο στόχο. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ναρκωτικών ε, και την ε, δυνατότητα που έχουν οι έμποροι ναρκωτικών ε, να προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση και να πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά από εμά. Και κάτι για τα φάρμακα. Δεν θέλουμε φυσικά να ελέγξουμε το σύνολο των φαρμάκων. Απλώς ε, θα υπάρχει μία εποπτεία ε, των φαρμάκων που είναι καταχωρημένα. Δεν ε, πρόκειται για εξαντλητικό εγχείρημα, αλλά δεν θα έπρεπε και πάλι στην έκθεση αυτή να χάσουμε τον κύριο στόχο. Τι θέλει η Ευρώπη στην πραγματικότητα. Θέλει να καταπολεμήσει τους ανθρώπους αυτούς ε, που διοχετεύουν ε, τις ουσίες αυτές, ε, καταχρώνται τις ουσίες αυτές για να τις χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή ναρκωτικών. Ωραία. κατά προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών σε μία εβδομάδα από σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα. Και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στην επόμενη τακτική μας συνεδρία στο Μάρτιο. Σας ευχαριστώ όλους. Σημείο 7. Okay. This... Uh, ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη Τομάς Μας εξ εξονόματος της Κωνσταρικάνης Προεδρίας του Συστήματος Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής. Να καλωσορίσω τον πρέσβη, τον Μας Δουένιας που εκπροσωπεί εδώ την Κωνσταρίκα γιατί είναι η χώρα που έχει την προσωρινή προεδρία του συστήματος ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής και να καλωσορίσουμε και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους από τους πρέσβη της Κεντρικής Αμερικής που βρίσκεται εδώ σήμερα. Ο πρεσβευτής Ντουένιας ήταν σημαντικός συνομιλητής μας για το ζήτημα της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής και συμμετείχε σε μία από τις δημόσιες ακροάσεις που υλοποιήσαμε πέρυσι για τις εμπορικές και οικονομικές προοπτικές των Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι ο κύριος ε, Σούλτς ε, συμπεριέλαβε την Κωνσταντίνα την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην ε, Λατινική Αμερική και επανέλαβε στην ομιλία του στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το στόχο να έχουμε στενότερες εμπορικέ σχέσεις με βασικούς εταίρους όπως είναι η Λατινική Αμερική που θεωρεί ζωτική για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν τον κύριο Πρέσβη να αναφερθεί συγκεκριμένα στα ζητήματα αυτά και στη διαδικασία ακύρωσης της συμφωνίας ε, με την Κεντρική Αμερική και την προετοιμασία για την ε, εφαρμογή των εμπορικών πτυχών της συμφωνίας. Γιατί αυτή δεν είναι, μόνο μια, δεν είναι μια συνθέτη συμφωνία, αφορά μόνο το εμπόριο. Και θα ήθελα να σας καλήσω να αναφερθείτε στα θέματα αυτά. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, καθηγητά Μορέιρα, για την ευγενική πρόσκληση που μας κάνατε ως πρόεδρο, προσωρινό πρόεδρο του Συστήματος Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής, του ΣΥΚΑ, για να αναφερθούμε στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που μας ε, περιμένουν ε, ε, μετά την ε, προσεχή ισχύ τη συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ημών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ και κυρίως τους βουλευτές Παύλο Ζάλβα και Γιώργ Λάιτφριντ ε, ως εισηγητής και της συμφωνίας και του κανονισμού εφαρμογής της ε, διμερούς ρήτρα ε, διαφύλαξης και του μηχανισμού σταθεροποίησης της μπανάνας για την Κεντρική Αμερική. Το έργο σας, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, είναι γνωστό και σας ευχαριστούμε ε, γι' αυτό. Οι πρέσβεις της Γουατεμάλας, του Σελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας, της Νικαράγουας, του Παναμά και φυσικά της χώρας μου, της Κωνσταντίνα. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία ακύρωσης στην Κεντρική Αμερική, ε, με χαρά σας ενημερώνω ότι όταν δόθηκε η έγκρισή μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκίνησε αμέσως η διαδικασία συζήτησης της συμφωνίας στις ε, νομοθετικές μας ε, συνελεύσεις στα κοινοβούλια μας και ταυτόχρονα ξεκίνησε η διαδικασία ε, καταγραφής των Ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων ε, που είναι προϋπόθεση για την ισχύ της συμφωνίας. Θα ήθελα λοιπόν με τα χαράς να σας ενημερώσω ότι δύο χώρες της περιοχής, η Νικαράγουα και η Ονδούρα, κύρωσαν τη συμφωνία και οι υπόλοιπε είναι στη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας και αυτό ε, είπαμε και στον πρόεδρο Σούλτς ε, κατά την επίσκεψή του στην Κεντρική Αμερική. Επίσης, η διαδικασία ε, συμπερίληψης των γεωγραφικών ενδείξεων έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε μια συνεδρίαση η οποία έγινε μεταξύ Υπουργών Εμπορίου Κεντρικής Αμερικής και του ε, Επιτρόπου Ντεγούχτ στα τέλη του περασμένου μηνός στο Σανδιάγο αποφασίστηκε να κάνουμε μία απόπειρα να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες μας ε, κύρωσης και γεωγραφικών ενδείξεων μέχρι τις 15 Μαΐου, ε, έτσι ώστε να δοθεί η προσωρινή εφαρμογή του εμπορικού τμήματος της Συμφωνίας ε, εντός του μηνός Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τι προόδου που έχουν γίνει σε θέματα ολοκλήρωση, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η έγκριση τη συμφωνία από το Κοινοβούλιο ε, δημιούργησε πολύ θετικές προσδοκίες ε, και υπήρξαν πολύ ε, σημαντικές πρόοδοι στο θέμα της ολοκλήρωσης. Καταρχάς, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι πρόεδροι των χωρών μας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον πρόεδρο Φαναρόμπαϊ, τον πρόεδρο Μπαρόζο και τον πρέσβη Λέφλερ, ο οποίος εκπροσωπούσε την Βαρόνη, Άστον, Άστον στο Σαντιάγο για να συζητήσουν δύο πολύ συγκεκριμένα θέματα την ασφάλεια και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Και εμφωνήθηκε να προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μας βοηθήσει για την διαδικασία η οποία ήδη είναι εξελίξη, για την θεσμική ενίσχυση του συστήματος ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής, που είναι μία από τις προτεραιότητες της προσωρινής Προεδρίας της Κωνσταντίνα. Ε, εχθές ε, στο Σαν Χωσέ, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Κωνσταντίνα, ο κ. Ενρίκε Καστίγιο, ε, εγγενίασε την πρώτη συνεδρίαση ε, συμβούλων του ΣΥΚΑ, στην οποία υπήρχε μια μερίτσια διάταξη που περιλάμβανε μια πρόταση της Προεδρίας της Κωνστανταρίκας για την ανανέωση και την ενίσχυση σε θεσμικό επίπεδο του ΣΥΚΑ και παρουσιάστηκαν μια σειρά από συγκεκριμένε προτάσεις προκειμένου να τροποποιηθούν τα βασικά περιφερειακά όργανα. Επίσης θα ήθελα ε, να σας ε, ε, ενημερώσω ότι και ο Παναμάς συμπεριλήφθηκε στο υποσύστημα οικονομικής ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής, το ΣΥΕΚΑ, και με αυτό ολοκληρώνεται η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση. Και τέλος, εξακολουθούν να έχουμε σημαντικές πρόοδους και διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην Κεντροαμερικανική Τελωνιακή Ένωση. Τι μελιγενέστε τώρα. Αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, προβλέπεται αύξηση στο διμερές εμπόριο. Φυσικά το ποσοστό θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν οι εισαγωγείς ή οι εξαγωγείς ε, εκατέρωθε. Αλλά πέραν της εμπορικής ροής ε, θα πρέπει να αναμένεται και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή, ε, με βάση βέβαια και την τόσο σημαντική αλλαγή που προβλέπει η συμφωνία που είναι η αντικατάσταση του συστήματος ε, SPG, το οποίο δεν βοηθούσε το κλίμα των επενδύσεων, ενώ αυτή τη στιγμή με την συμφωνία ε, βοηθάτε. Η συμφωνία θα μας βοηθήσει επίσης να ε, ανταλλάξουμε γνώσεις, τεχνολογία και καινοτομία και θα μας εκθέσει στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Από πλευράς μας οι νέοι μας εταίροι θα μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην περιφερειακή μας αγορά, καθώς και μια ανταγωνιστική πλατφόρμα παραγωγής ε, αγαθών και υπηρεσιών. Ε, επειδή υπάρχει μια περιοχή με 40 εκατομμύρια κατοίκους που επιθυμούν να παράγουν και να είναι ανταγωνιστικοί, ε, θα ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πρόκειται για μια περιοχή η οποία προσβλέπει στην ένταξή της στον νόσα και επίσης έχουμε και μια υποψήφια χώρα στην Γενική Διεύθυνση του, του ΠΟΕ στη συμφωνία υπάρχει λοιπόν και ένας πυλώνας συνεργασίας, ο οποίος ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο συγκεκριμένα στην ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, όπως ε, ε, το λέμε στα αγγλικά capacity building. Μόνο έτσι, μαθαίνοντας τις καλύτερες τεχνικές, θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με βιώσιμο τρόπο και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολιτών μας. Αυτός είναι ο πραγματικός άλλωστε σκοπός της συμφωνίας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. OCDE Η είναι υποψήφη για την ένταξη στον ΩΣΑ, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωσή σας σχετικά με την ε, επικυρώση της συμφωνίας αλλά και με την περιφερειακή ολοκλήρωση στην Λατινική και την Κεντρική Αμερική. Ας προχωρήσουμε τώρα στα μέλη της Επιστροπής. Αρχίζουμε με τον ε, Πάμπλο. Αναγνωρίζετε, πιστεύω, την, ε, τον όγκο της δουλειάς που έχει κάνει αυτή η Επιτροπή και ο εισηγητής, ο κύριος Τάου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα βιανικά σας λόγια. Να καλωσορίσω και τον ε, κύριο Πρέσβη και να τον ευχαριστήσω για τα όσα είπε ήταν ε, μεγάλη τιμή να συνεργαστούμε μαζί του και μαζί με τους συναδέλφους και τους κοιόδες συζητητές και με τη βοήθεια του Πρόεδρου και την Γραμματεία. Καταφέραμε κάτι, όχι εύκολο. Σε αυτό τον οίκο όμως ε, μπορώ να σας πω ότι η αποστολή εξετελέστη. Εγώ χαίρομαι πολύ για τα όσα μας είπε ο κύριος Πρέσβης, για τις γεωγραφικές ενδειξίες, για την κυρίωση από την Ονδούρα και την Ικαράγουα. Ε, μακάρι να έχουμε πιο θετικά νέα και μακάρι η πρόβλεψή σας ε, να βγει αληθινή, δηλαδή την 1η Ιουνίου να είναι τεθεί προσωρινά σε ισχύ ε, το εμπορικό τμήμα της συμφωνίας. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν μια χρυσή εποχή είναι μια ιστορική ευκαιρία αυτή η συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Κεντρική Αμερική, όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης, για να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και νομίζω ότι αυτό εκπροσωπεί η χώρα σας και η παρουσίαση της σήμερα αποτελεί ε, μια ευκαιρία για την ανάπτυξη χώρας της Κεντρικής Αμερικής ε, και για πρόθεση της κοινωνικής συνοχής και αποτελεί και μια ευκαιρία για πρόθεση της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Κεντρική Αμερική. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα έχει μια δυναμική αυτή συμφωνία που δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη και μακάρι το συντομότερο δυνατόν και η Κεντρική Αμερική αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν να κατανοούν ποια είναι τα ωφέλη και αυτά τα ωφέλη να κατευθυνθούν κυρίως προς τους πολίτες. Και εγώ πιστεύω ότι δεν συμβαίνουν τυχαία τα πράγματα και όπως είπε και ο Πρόεδρος Μορέιρα, η Κώστα Παρουσίαση υποψηφιότητα ε, για ε, πρόεδρο του ΠΟΕ. Ε, ποτέ νομίζω ένας Λατινοαμερικανός δεν ήταν πρόεδρος του ΠΟΕ, έτσι λοιπόν ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε δυο λόγια για το πώς βλέπετε ίσως αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Πρέσβη. Ευχαριστώ Παμπλό. Είμαι σίγουρη ότι σίγουρος ότι και οι επόμενοι συνάδελφοι θα καλωσορίσουν τον καλεσμένο μας ε, ακόμα και όσοι λείπουν. Η επόμενη η Φραντσίσκα Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε καταρχάς. Έχω πολλές ερωτήσεις, θα περιοριστώ όμως σε ορισμένες. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα σχετικά με το πώς ακριβώς η εμπορική διάσταση θα εφαρμοστεί στην Κεντρική Αμερική, ιδιαίτερα ε, εφόσον υπάρχουν διαφορές στην διαδικασία επικύρωσης, για παράδειγμα για τις ποσοστώσεις, τι θα γίνει. Θα χρησιμοποιηθούν ε, με την αρχή του όποιος έρθει πρώτος ή όλες οι χώρες, ή αφότου όλες οι χώρες επικυρώσουν τη συμφωνία. Επίσης, Φαντάζομαι πως έχετε ήδη δει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις σχέσεις με την Χιλή και το Μεξικό, τα καλά και τα άσχημα και αναρωτιέμαι πώς θα αντιμετωπίσετε ζητήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί ως ελλείψεις από τις προηγούμενες συμφωνίες, δηλαδή τις αυξημένες ανισορροπίες στο εμπόριο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την έλλειψη διαφοροποιημένων εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αφόσον ολοκληρωθούν αυτές οι συμφωνίες, τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά που αυξάνονται. Πώς ε, σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά στην Κεντρική Αμερική έτσι ώστε να μην επαναληφθούν. Επίσης, γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στόχαστρο λόγω της ε, φοροδιαφυγής στην Λατινική Αμερική και στην ε, διαφορετική τιμολόγηση η οποία πρακτική έχει κοστίσει πολύ στους ε, εθνικούς προϋπολογισμούς. Και το κεφάλαιο με τις, που αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μάλιστα προβλέπει κάποιες να νομιμοποιηθούν. Εσείς πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε στην Κεντρική Αμερική έτσι ώστε να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή και να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον πρέσβη για τα καλά του λόγια του και για την εισαγωγή του. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις ε, συζητήσεις με θέματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής. Ε, αρχίζοντας με την έκθεση πρωτοβουλίας που συνέταξα για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής, ασχολήθηκα με το πώς ακριβώς η συμφωνία αυτή προωθεί τη συνεργασία και το εμπόριο ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ποια προγράμματα και ποιες πρωτοβουλίες χρειάζονται για να στηρίξουν περαιτέρω την συμφωνία σύνδεσης που να ωφελούν και τους πολίτες. Στάθηκα σε ένα σχολείο σας όπου είπατε ότι ένα από τα... Ένας από τους στόχους σας είναι η συμφωνία αυτή να προωθήσει την βελτίωση της, ε, των συνθήκων ζωής των πολιτών στις χώρες σας. Αυτό σημαίνει δηλαδή την προστασία των τοπικών επιχειρήσεων από πιθανές απειλές που έχουν ε, άμεση σχέση με τη Συμφωνία σύνδεσης επίσης ποια είναι τα νέα προϊόντα που σκοπεύετε να εξάγετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αυξήσετε και την ανταγωνιστικότητα της περιφερειάς σα, πέρα από αυτά που ήδη υπήρχαν στην προηγούμενη συμφωνία. Επίσης, κάτι παρόμοιο με αυτό που είπε και η συνάδελφος Φραντσίσκα Κέλλερ σχετικά με τις επενδύσεις και την εφορολόγηση του εμπορίου και τα προβλήματα που αυτές έχουν. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για παράδειγμα, έγινε μία μελέτη από μία Ολλανδική ΜΚΟ που έδειξε τις ε, σχέσεις οι οποίες καθιστούν μία απειλή και μια δυναμία ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγξει το ξέπλυμα χρήματος και την φοροαποφυγή. Πώς σκοπεύετε εσείς να το αντιμετωπίσετε, να το ελέγξετε και να το αποτρέψετε. Ποια είναι το πρόγραμμά σας. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω βασισμένη στις ε, σχέσεις ε, με τη Χιλή και το Μεξικό και βασισμένη στην ε, εκτίμηση αντικτύπου για, τις, για τη συνεισφορά της συμφωνίας αυτής στην η οικονομική δυνατότητα της Χιλής να αναγνωριστεί ως πλήρης εμπορικός εταίρος. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν για τα αποτελέσματα. Αν αυτά ήταν σαφή ή όχι. Θα, σύμφωνα με την πελέτη θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε αυτό με κάτι θετικό, αλλά δεν είναι προφανές αυτό. Δεν είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα της συμφωνίας είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις περιπτώσεων όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε στο Μεξικό και τις συνέπειες για την ασφάλεια των τροφίμων, για το μέλλον των ε, μικρών και μεσαίων αγροτών που παράγουν για παράδειγμα φασόλια και ρύζι, για την ε, έκταση των, ε, της μονοκαλλιέργειας στη χώρα σας για παράδειγμα την καλλιέργεια του ανανά και το πώς αύξηση, η πίεση για την αύξηση της ε, ζήτησης επηρεάζει την γεωργία και τι σημαίνει αυτό και για τους αγρότες. Και τέλος, η ολοκλήρωση της ε, συμφωνίας αντιμετωπίστηκε με κάποια κριτική διάθεση από τους ε, συνδικαλιστές της χώρας σας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τώρα πώς θα συμπεριλάβετε αυτή την κριτική στις προσπάθειές σας να ξεπεράσετε τις ανησυχίες που διατύπωσαν εκείνοι και να τους δείξετε ότι το πρόγραμμά σας είναι ολοκληρωμένο και θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων που βρίσκονται στη συμφωνία που υπογράψατε. Ευχαριστώ πολύ. Μαριάν Σαρνές τώρα από την ομάδα Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτά προς την πλευρά της Λατινικής Αμερικής. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Καλό είναι που το πράττει. Ήμουν στο Σαντιάγο στη Χιλή για τη Σύνοδο Κορφής Γιουρολάτ πριν δύο-τρεις εβδομάδες όπου 33 χώρες της Λατινικής Αμερικής έλαβαν ε, μέρος και με ξέπληξαν ε, δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, η ΣΥΚΑ, η Μερκοσούρ, ε, υπάρχει και ένας αριθμός χωρών που έχουν μπει σε μία ένωση ε, μαζί με τη Χιλή και πρόκειται για χώρες ε, που ε, βρίσκονται στον Ελληνικό ωκεανό. Εσείς οι χώρες Κεντρικής Αμερικής έχετε κατά νου να οργανωθείτε με πολιτικό τρόπο όπως αυτές τις 33 χώρες ή θα συνεχίσετε να συνεδρίσετε σε διαφορετικούς οργανισμούς. Δεν ε, ξέρω αν ε, πρέπει να συνεδριαστεί όχι Χελά σε αυτή την σύνοδο ε, με τη Λατινική Αμερική, Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τρει χώρε ήταν εκεί και ήταν χρήσιμο. Και κάτι ακόμα που άκουσα στη Χίλη από την ευρωπαϊκή πλευρά. Άκουσα δύο μεγάλες ανησυχίες. Πρώτη ανησυχία για τον προστατευτισμό μια σειρά χωρών, ιδίως της Αργεντινής, για να μην την κατανομάσω. Ε, και κυρίως την ανησυχία αυτή την έχουν οι Ευρωπαίοι αλλά όλοι και όσοι βρίσκονται στη Λατινική Αμερική που δεν μπορούν να εσώτιμους όρους ε, να προβούν σε εμπόριο επίσης την εγγύηση για τις ξένες επενδύσεις ιδίως στις ευρωπαϊκές ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου δεν είναι καθόλου σταθερό το νομικό πλαίσιο και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τις επενδύσεις αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό και τρίτη ανησυχία προερχόταν από κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και φορούσε την, το άνοιγμα στην αγορά και μια μεγαλύτερη πίεση που ασκείται στους φυσικούς πόρους, κυρίως τα ορυκτά. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου κύριε Πρέσβη και σας ευχαριστώ για την απάντησή σας εκ των προτέρων. Πρόεδρος ε, και τέλος ε, Κλάσφιτ ε, που έφτασε τώρα τελευταία, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ήδη ενημερωθεί για την ομιλία του προσκεκλημένου μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Λυπάμαι πολύ που άργησα. Αλλά σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη και πολλές συνεδριάσεις. Χαίρομαι όμως που κατάφερα να έρθω. Και ο κύριος Λάγκε με ενημέρωσε πλήρως για όσα ελέγχθησαν. Και είμαι απόλυτα λοιπόν ενημερωμένος, Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις έχω. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την εμπορική συμφωνία, διότι ήμουν και ο εισηγητής για τις ε, ρήτρες διασφάλισης για την ε, Κεντρική Αμερική και ο σκιώδης εισηγητής για την ίδια την έκθεση. Ε, έχω να ρωτήσω. Η ρήτρα διασφάλισης είναι λίγο πολύ προορισμένη για να προστατεύσει την ε, βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει και ε, κάποιες ε, επιρροές στην καλλιέργεια μπανάνα στην Κεντρική Αμερική. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω το πώς εκτιμάτε εσείς ότι θα λειτουργήσει αυτό σε πραγματικές συνθήκες. Αναμένετε προβλήματα με αυτή τη ρήτρα διασφάλισης εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν προβλήματα ή θα γίνει αυτό, αλλά έπειτα, νομίζω πως οι συνάδελφοι ήδη το ανέφεραν, όμως θα ήθελα και εγώ να το ρωτήσω. Τι γνώμη έχετε για την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνδέσει τα εμπορικά ζητήματα με άλλα, για παράδειγμα με κοινωνικά ζητήματα ή με περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό και θα ήθελα να γνωρίζω και την άποψη των εταίρων μας γι' αυτό. Έπειτα, κάτι τελείως διαφορετικό, που δεν έχει σχέση με το εμπόριο, αλλά με διπλωματική πολιτική. Βρέθηκα στην ε, συνάντηση στην ε, Χιλή ως μέρος της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας λίγες εβδομάδες πριν και αναφέρθηκε στα πλαίσια των συζητήσεων ότι δεν βοηθάει όταν μία πλευρά μπλοκάρει ουσιαστικά τα πράγματα. Στην περίπτωση αυτή υπήρχε μία ξεχωριστή ψηφοφορία και όταν η μία πλευρά ψηφίζει κατά, η άλλη πλευρά δεν μπορεί να αντιδράσει. Θα με ενδιαφέρε λοιπόν να μάθω τις απόψεις της ε, λατινοαμερικανικής πλευράς για το θέμα αυτό, διότι έχω διαπιστώσει ότι πολλές φορές εμείς, η ευρωπαϊκή πλευρά, έχουμε μπλοκάρει θέματα τα οποία είναι προς όφελος και αντικατοπρίζουν τα συμφέροντα της ε, κεντρικής Λατινικής Αμερικής, τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα. Thank Σας ευχαριστώ. Και τέλος να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ματίας Γιώργηρσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνω κάποια σύντομα σχόλια και από τη δική μας πλευρά σε σχέση με όσα παρουσίασε ο κ. Πρέσβης. Συμφωνείτε με την αισιοδοξία του με την αισιοδοξία απόψή του. Καλώς ορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαδικασία της κύρωσης και από τις δύο πλευρές. Και νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δυναμική και βούληση στην Κεντρική Αμερική για να προχωρήσουν γρήγορα. Έχουμε θέσει μία ημερομηνία στο Σαντιάγο στις 15 ε, Μαΐου να είναι έτοιμη η Κεντρική Αμερική να έχουν πληρωθεί όλες ε, οι εσωτερικέ διαδικασίες για την κύρωση και να έχουν εκπληρωθεί και όλα όσα πρέπει να γίνουν στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων και στο τομέα της ε, διαδικασίας καταχώρησης και στον τομέα της νομοθεσίας. Πολλά πρέπει να γίνουν από την πλευρά τη Κεντρική Αμερική, αλλά νομίζω υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση και αυτό είναι σημαντικό. Εμεί, από την πλευρά τη Κομισιόν συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους εταίρους από την Κεντρική Αμερική και ήδη έχουμε τις διαδικασίες καταχώρησης να προχωρούν ομαλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπάρχει προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Και αν γίνει επαρκής πρόοδος, την 1η Ιουνίου, η 1η Ιουνίου ακούγεται σε μια ρελιστική ημερομηνία, όπου ελπίζουμε όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής να είναι σε θέση να μπορέσουν να εφαρμόσουν προσωρινά τη συμφωνία. Αυτή είναι η συνολική μου αξιολόγηση για την κατάσταση. Έχει γίνει πρόοδος, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε δουλειά ενώπιόν μας. Από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζουμε, η Κομισιόν δηλαδή, ελπίζει να υπάρξει πρόοδος στη διαδικασία κύρωσης. Όχι μόνο στην Κεντρική Αμερική, αλλά και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά πρέπει να κυρώσουν τη συμφωνία. Ε, νομίζω ότι μόνο τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε το εμπορικό τμήμα της συμφωνία. Για να το κάνουμε αυτό όμως ε, θα πρέπει να τεθεί όλη η σύμφωνη σε ισχύ. Υπάρχει και σημαντική πτυχή συνεργασίας. φέρθηκαν κάποιοι βουλευτές σε αυτό, πώς ε, συνδέουμε το πολιτικό κεφάλαιο με το κεφάλαιο της συνεργασία, με το εμπορικό κεφάλαιο. Όσο γρηγορότερα τεθεί σε ισχύ όλη η συμφωνία, τόσο ταχύτερα θα έχουμε ένα διάλογο και μια ευρεία συνεργασία με την Κεντρική Αμερική. Αν μου επιτρέπετε, να κάνω και κάποια σύντομα σχόλια για όσα υπόθηκαν. Για τους ΕΛΑΚ. Για μας ε, ήταν επιτυχής η Σύνοδος Κορφής. Ήταν ε, ενδιαφέρον ε, να βλέπουμε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση και διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών Λατινικής Αμερικής Καραϊβικής. Ήταν και συνάντηση όχι μόνο κυβερνήσεων, αλλά και μεταξύ βουλευτών. Είχαμε και μια δικαστική σύνοδο κορφής Είχαμε δηλαδή ψηλό επίπεδο συμμετοχή και από Ευρωπαίου ηγέτε. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η δήλωση που προέκυψε. Ισχυρή πολιτική υποστήριξη για πιο στενούς δεσμούς. Φυσικά είναι διπλό το ενδιαφέρον και από τη Λατινική Αμερική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε όλο ένα και μεγαλύτεροι εταίροι. Αυτό είναι καλό στείλαμε ισχυρό μήνυμα κατά του προστατευτισμού στην δήλωση της Συνόδου Κορφής. Επίσης, ε, στείλαμε το μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα και είπαμε, αν δείτε τη δήλωση και συγκεκριμένα την παράγραφο 21, θέσαμε μία σειρά στόχων για όλες τις διαδικασίες που έχουμε με τις υπομάδες στη Λατινική Αμερική. Συνολικά λοιπόν ήταν πολύ καλή η Σύνοδος Κορφής και χρησιμοποίησαμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ μιας επίσημης συνάντησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της συνάντησης του Επιτρόπου Ντεγκούχτ και των εταίρων του. Πώς μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη συμφωνία. είναι αρκετά τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα κυρώσει. Δεν έχω τον κατάλογο και τον 27. Δεν είπαμε να τους ε, εξευτελίσουμε, απλώς να μας πείτε ποιοι είναι. Ε, θα επανέλθω και θα σας απαντήσω. Κύριε Πρέσβη, αρκετά σχόλια, αρκετές ερωτήσεις, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να απαντήσω στον φίλο μας τον Παύλο Σάλβα στη μητρική του γλώσσα και θα προσπαθήσω για λόγους ευγένειας να απαντήσω και στους υπολείπους ε, στα αγγλικά. Ελπίζω να τα καταφέρω και τα δύο ταυτόχρονα. Καταρχάς, τον ε, Παύλο, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για όλα όσα έχετε κάνετε και εσείς και ο κύριος Λάιτφιριτ ε, για την περιοχή μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα μαζί σας διότι μας ανοίξατε την πόρτα για μια ιστορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι το αντιμετωπίζουμε εμείς. Η Κωνσταντίνα, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, είναι υποψήφια για την ε, διεύθυνση του ΠΟΕ. Είναι νέα υποψήφιες χώρες αυτή τη στιγμή και μετά από μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε ε, πρόσφατα ε, δόθηκε ε, χώρος σε κάθε έναν από τις υποψήφιες χώρες να κάνουν τις παρουσιάσεις τους και από εκεί και πέρα υπήρξε και μια συνέντευξη τύπου. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι γυρίζουν τον κόσμο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και παρουσιάζουν τη διαπιστευτήριά τους και ελπίζουμε ότι ε, η διαδικασία που ξεκίνησε στη Γενέβη να μας οδηγεί σε μια τελική επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που τα αναφέρετε. Η Κωνσταντίνα έχει αυτή τη φιλοδεξία. Πιστεύει ότι μια μικρή χώρα μπορεί να είναι ε, ένας καλός συνεργάτης ε, στον ΠΟΕ και θα προσπαθήσει να είναι διαμεσολαβητής ε, σε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο διεθνές εμπόριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που τα αναφέρετε. Η κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και θα ήθελα να πω και ιδιαίτερως για το ενδιαφέρον σας. Στις συζητήσεις που κάναμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, διότι είμαι εδώ, εδώ και δύο χρόνια, ε, κατέστη ότι το νόημα αυτής της σχέσης με την Ευρώπη είναι μακρόπνο, διότι θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο και πολύ πιο μακρινό από μια εμπορική συμφωνία. Θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήμασταν ιδιαίτερα τυχεροί που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει μια συμφωνία σύνδεσης, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο συμφωνία που μπορεί να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπερ και σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο ένα πεδίο εφαρμογής για το τωρινό και το μελλοντικό εμπόριο και τους κανόνες που θα διέπουν το εμπόριο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι και κοινωνικά και ε, αποδεκτές ε, εμπορικές πρακτικές. Αλλά υπάρχει και μία συνεργασία που είναι σημαντική, διότι πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητες και να ενισχύσουμε τους θεσμούς της περιοχής μας, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να προβάλλουμε τις προτάσεις και τις πολιτικές που χρειάζονται για την ανάπτυξη των λαών μας. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μία βάση πολιτικού διαλόγου, που είναι εξίσου σημαντικό, ε, διότι μας προσφέρει μία πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χώρες μας, οι ηγέτες μας και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουν να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσουν ειλικρινά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται λοιπόν για μια συνολική συμφωνία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από το εμπόριο και το να το βλέπουμε μόνο από την οπτική γωνία του εμπορίου είναι άδικο. Διότι αυτό το οποίο επιθυμούμε και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και η ραχοκοκαλιά αυτής της συμφωνίας είναι θεσμική μεταρρύθμιση, ενίσχυση του κράτους δικαίου, προστασία των δικαιωμάτων των ε, ε, αδυνάμων και μία απόπειρα να δημιουργήσουμε και να μάθουμε πώς να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε καλύτερα μέλη ε, της κοινωνικής, οικονομικής και εργασιακής κοινότητας. Πρόκειται λοιπόν για μία συνολική προσέγγιση, αν θέλετε. Και όπως γνωρίζετε, μια συμφωνία σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό λοιπόν το οποίο επιθυμούμε είναι μέσω αυτών των διεθνών δεσμεύσεων, διότι δεν πρόκειται απλώς για δέσμευση της Κεντρικής Αμερικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ε, αναλάβει και αντίστοιχε δεσμεύσει και με τι Ηνωμένες με τον Καναδά, το Μεξικό, ε, την ε, Καραϊβική, η Κωνσταντίνα έχει μια συμφωνία και με την Κίνα ε, με τη Σιγκαπούρη, με τη Χιλή. Συνεπώς λοιπόν, στη διάρκεια των προσπαθειών της Κεντρικής Αμερικής, δημιουργούμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία σχέση με τον κόσμο η οποία ου μόνον θα μας κατευθύνει και θα μας συνδράμει για να έχουμε προτιμησιακή πρόσβαση, αλλά θα μας διδάξει και πώς θα είμαστε καλύτεροι στις κοινωνίες μας. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό απαντά σε κάποιες από τις ανησυχίες σας, διασκεδάζει κάποιες από τις ανησυχίες σας και ε, επαναλαμβάνω ότι η ραχογοκαλιά είναι το κράτος δικαίου. Όλοι θα πρέπει να πληρώνουν ίδιους φόρους, όλοι θα πρέπει να τηρούν τις ίδιους κανόνες και αυτό επιθυμούμε εμείς στην περιφέρειά μας. Και φυσικά εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, θα προσέχετε ε, ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Κύριε Σόλτς, χαίρομαι ιδιαίτερα ε, κάθε φορά που σας ακούω. Και πάλι εκτιμώ ιδιαίτερα τα καλά σας λόγια. Αναφερθήκατε στο κατά πόσον θεωρούμε ότι υπάρχει επαρκή στήριξη για αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι υπάρχει. Φρονώ ότι είναι ένα καλό εφαλτήριο. Οι συμφωνίες αυτές είναι ζωντανές ε, αν μου επιτρέπεται όρος, προσφέρουν τη δυνατότητα αλλαγών μέσω πολιτικού διαλόγου, μέσω συναντήσεων, μέσω επιτροπών και ούτω καθεξής και επομένως μπορούν να γίνουν ένας πολύ επικοδομητικός τρόπος ε, αλληλεπίδρασης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, περίπου ο νονός της περιοχής. Πριν από πάνω από 20 χρόνια μας βοηθήσατε ε, σε πολύ χαλεπούς καιρούς ε, και πολιτικούς και κοινωνικούς. Και η ΣΥΚΑ, η Συμφωνία Ολοκλήρωσης Κεντρικής Αμερικής, για να επανέλθω και σε μία ερώτηση για το θεσμικό ρόλο, η ΣΥΚΑ λοιπόν είναι το αρχαιότερο σύστημα της Λατινικής Αμερικής. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής είναι η μόνη ολοκληρωμένη περιοχή στη Λατινική Αμερική. Μπορεί να είμαστε μικρές χώρες και να μας πήρε μεν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αναζητούμε συνεχώς πώς θα γίνουμε μια ισχυρότερη περιοχή, με όλες βέβαια τις δυσκολίες που συμπεριλαμβάνει κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν που αναζητούμε και συνειδητοποιούμε ε, είναι ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από το εμπόριο. Και πάλι αφορά θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας και δεσμεύσεις ε, των πολιτικών μας κομμάτων για τη θεσμική μεταρρύθμιση. Κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και εσείς γνωρίζετε ως νομοθέτες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχουμε σε τοπικό επίπεδο ε, θεσμική μεταρρύθμιση. Είναι πόδινο. Ε, μέσω των διεθνών μας δεσμεύσεων αρχίσαμε να οικοδομούμε σιγά σιγά μια ισχυρή θεσμική δομή στην ε, ε, Κεντρική Αμερική και η Κώστα Ρίκα τώρα αναζητά με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πρόεδρε, να μεταρρυθμίσουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να μας βοηθήσετε στο σχεδιασμό ενός ε, σύγχρονου, διάφανου και αποτελεσματικού θεσμού που θα εκπροσωπεί την περιοχή μας. Και τέλο, για να ολοκληρώσω, ο κύριο Σόλτ, βεβαίως και μας ανασυχεί το θέμα της ασφάλειας. Η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο γνωρίζει σαφέστατα η περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και τα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη μεταξύ της ε, Προεδρίας μας και της Προεδρίας των δικών σας θεσμικών οργάνων ήταν ε, τα εξής. Το ένα ήταν η ασφάλεια ε, που αφορά τη νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, την ε, ε, πορεία ναρκωτικών, παράνομη μετανάστευση και το καθεξής, καθώς επίσης και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες της περιοχής. Η κυρία Τεσσαρνέ. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είναι πολλοί οι θεσμοί που εκπροσωπούν διάφορες ομάδες χωρών στη Λατινική Αμερική. Και αυτό ε, αποτελεί συνεχή μας ανησυχία. Ωστόσο, θα ήθελα να περιοριστώ στη ΣΥΚΑ, στο Σύστημα Ολοκλήρωση τη Κεντρική Αμερική, διότι εμεί ε, εκπροσωπούμαστε εκεί, από τη Γουατεμάλα μέχρι τον Παναμά, ε, και υπάρχουν και μία σειρά από άλλε οργανώσει. Αλλά αυτό το οποίο αναζητούμε είναι με τη βοήθειά σας να δημιουργήσουμε έναν ισχυρότερο θεσμό, ο οποίος θα είναι πιο σύγχρονος, πιο διάφανος και θα μας βοηθήσει να ε, καθοδηγήσουμε τις κυβερνήσεις μας και την περιοχή μας σε καλύτερες εποχές, με τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι αρκετές οι προκλήσεις ε, για την περιοχή μας. Σημειώνω βεβαίω αυτά που μας είπατε και δεσμευόμαστε για μια ισχυρότερη ολοκλήρωση στην περιοχή μας. Ο κύριος Λάιτφριτ, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι για την ε, δυνατότητα αυτή που μου δίνετε. Θέσατε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν νομίζω βέβαια ότι έχω μια σωστή απάντηση να σας δώσω, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια απόπειρα να σας δώσω μια εικόνα. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριέ μου, η ρήτρα διασφάλισης ε, ήταν ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Ήταν μια ιδιαίτερη διαπραγμάτευση και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός αυτός, διότι το θέμα της μπανάνας ήταν διαφιλονικούμενο ε, για σχεδόν ένα 25 ε, χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα. Και η ανησυχία αυτή της Ευρώπης ιδίω διασκεδάστηκε από αυτή τη νομοθεσία για τη ρήτρα διασφάλισης. Αναμένουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, διότι γνωρίζουμε πόσο εις βάθος έχει πάει η συζήτηση, πόσο έχει προχωρήσει η συζήτηση και δεν νομίζω ότι είναι πολλές οι χώρες που είναι διατεθειμένες να θέσουν το θέμα επιτάπητος και πάλι. Ελπίζω λοιπόν να ε, είστε καθησυχασμένος και να πιστέψετε ότι αυτή η ρήτρα διασφάλισης είναι ασφαλής. Και πάλι σας ανησυχεί το κατά πόσον υπάρχουν και τα κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω ότι προσπάθησα να είμαι σαφής. Είναι απόλυτη η δέσμευσή μας, διότι οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας, οποιαδήποτε μορφή εμπορίου, οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, οποιαδήποτε μορφή βιομηχανίας, έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατάσταση του λαού μας. Και αυτό το συνειδητοποιούμε απόλυτα και ελπίζω ότι με αυτή τη συμφωνία, και πάλι για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, θα υπάρξει μια νέα ε, σειρά ευκαιριών και προσβλέπουμε σε αυτές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, thank you, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιτρέψτε μου δύο σχόλια. Να πω καταρχάς πως για μένα όταν μια συμφωνία είναι καλή για τους εταίρους μας, είναι και στο χέρι τους να την αξιολογήσουν και πως τα... οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι το μόνο μέσο αξιολόγησης μιας συμφωνίας και του πόσο καλή είναι αυτή. Έπειτα, Όσον αφορά τους... την υποψήφια για την ε, θέση της ε, Γενικής Διευθύντριας του ΠΟΕ, όπως ε, σας ανέφερα, σας ανέφερα μία λοιπόν από του υποψηφίου είναι μια γυναίκα από την Κωνσταντίνα. Είναι πολύ ισχυρή η υποψηφιότητά τη. Θα ήθελα να με ενημερώσω λοιπόν και το κοινό και τα μέλη τη Επιτροπή για το ότι καταρχά υπήρχαν αρκετοί υποψήφοι που ζήτησαν να συναντηθούν μαζί μου και να μου παρουσιάσουν τι απόψει του και τις προσδοκίες τους για τον ΠΟΕ. Δέχτηκα να συναντηθώ μαζί του. Δεν θα αναφέρω φυσικά τα ονόματά του, Έπειτα, να πω ότι αυτή η Επιτροπή θα έπρεπε να ασχοληθεί ενεργά με την ε, διαδικασία αυτή και να τη συζητήσει εσωτερικά. Και θα προτείνω στην, ε, συζήτηση, στην συνάντηση των ε, συντονιστών τις απόψεις μου και πριν λοιπόν τη λήξη αυτής της διαδικασίας, την ολοκλήρωσή της, θα έχουμε και την δική μας συζήτηση για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εμείς θα πρέπει να ενεργήσουμε, μια που είμαστε και ο πιο σημαντικός εμπορικός ε, εταίρος στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Πιστεύω πως ε, ο ρόλος μας τον ΠΟΕ πρέπει να τονιστεί λοιπόν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτού του σημείου της ημερησίας διάταξης. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον πρέσβη της ε, Κωνσταντίνα, τον Μασδουένιας, αλλά και τους ε, πρέσβεις των ε, άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, της Γουατεμάλα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρα και του Παναμά. Σας ευχαριστώ όλους. Εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του σημείου αυτού. Σημείο 8. Ας αποχαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας, καταρχάς. Uh, Σημείο 8. Δραστηριότητες της εποπτικής ομάδας. Έχουμε αρκετές εποπτικές ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με τις εμπορικές μας σχέσεις με τους εμπορικούς μας εταίρους. Πρόσφατα οι ομάδες για την Ταϊβάν, Ινδία, Ρωσία και την Χιλή συνεδρίασαν και θα ακούσουμε τα αποτελέσματα τώρα των ε, συναντήσεών τους. Ας αρχίσουμε με τη Χιλή. Η ε, κυρία Κορέα Θαμόρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να σας ενημερώσω ότι στις 18 Δεκεμβρίου είχαμε την ομάδα για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής. Καταρχήν είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον Ματίας Γιώργενσεν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος μας έκανε μια σύντομη αξιολόγηση της συμφωνίας αυτής από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το 2003 Μέχρι φέτος 10 έτη λοιπόν ισχύει αυτή η συμφωνία και χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των εμπορικών ε, σχέσεων σε διμερές επίπεδο και των επενδύσεων. Ως ε, προς τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε αυτές τις εμπορικές σχέσεις, η Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι σε περιοδικές ε, συναντήσεις με τους εκπροσώπους και των δύο μέρων φάνηκε η βούληση και των δύο να εμβαθύνουν ε, στο εμπορικό, στην εμπορική πτυχή, όμως μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί μια ισορροπία συμφερόντων. Έχοντας ε, κατά νου και τη ρήτρα εξέλιξη, ε, που συμπεριλαμβάνεται στο εμπορικό κεφάλαιο της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής, η οποία θα επέτρεπε να προχωρήσουμε προς μεγαλύτερη απελευθέρωση. Σε τομεακό επίπεδο ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις το 2006 διαπραγματεύσεις που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Κομισιόν είναι ότι η αποτυχία στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, θα μπορούσε να οφείλεται κυρίως ε, στην απλωστομιακή διάσταση της εξελικτικής ρήτρα, ε, κάτι που δυσκολεύει την επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων. Η Κομισιόν έθεσε τη δυνατότητα να εστιάσει αλλού με ένα πιθανό καθολικό εξυγχρονισμό της συμφωνίας αυτής, τη ισχύουσα συμφωνίας σύνδεση που σας υπέσχε από το 2003 και κάτι τέτοιο θα μας διευκολύνει να συμπεριλάβουμε και ε, θέματα που δεν καλύπτονται μέχρι τώρα από τη συμφωνία αυτή σε ό,τι αφορά τους ε, γυμνούς εκπρόσωπου να σας πω ότι ο σύμβουλος ε, στο Υπουργείο Οικονομικών ε, δήλωσε την ικανοποίησή του για την αύξηση των διμερών της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και μας είπε ότι η Χιλή αυτή τη στιγμή σημειώνει σημαντική ανάπτυξη με χαμηλά ποσοστά ανεργίας παρά το ότι ζούμε σε εποχές κρίσης. Ε, ο χιλίος εκπρόσωπος ε, μας έδειξε ότι είναι πλήρως διαθέσιμος ε, να βρει μια ισορροπημένη λύση που να ωφελεί και τα δύο μέρη και επίσης ε, κλήθηκε να συμμετέχει σε συνεδρίαση στη Χιλή στο Σαντιάγο για να παρουσιάσει μια ομιλία σε σχέση με την προοπτική εξυγχρονισμού της συμφωνίας αυτής. Ε, σε ε, αυτή την ομιλία πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα να προχωρήσουμε προς μια καθολική και βάθος αναθεώρησης αυτής της συμφωνίας πέρα από το τομεακή εστίαση επίσης δεσμεύτηκα στην Επιτροπή να συνεχίσω να εργάζομαι στην ομάδα παρακολούθησης και να συνεχίσω να συνεδριάζομαι με εκπροσώπους της Κομισιόν όπως και εκπροσώπους της κυβέρνησης της Χιλής για να βρεθεί αυτή η ισορροπία συμφερόντων και να δούμε με ποιον τρόπο και με ποια μέσα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας αυτής. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε πιθανέ ημερομηνίε για πιθανή συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σας πιστεύετε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την της εμπορικής συμφωνίας. Δηλαδή για να υπάρχει εμβάθυνση μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την επιτροπή που έλαβε χώρα στη Χιλή. Υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα από τη χιλιανή κυβέρνηση να προχωρήσουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα δεύτερο στάδιο και πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε για να εμβαθύνουμε τις σχέσεις αυτές. Το θεμελιώδη στοιχείο που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, νομίζω υπόθηκε και από την Κομισιόν σήμερα το πρωί, είναι αυτή η πολιτική ενεργοποίηση και η πολιτική βούληση που έχει εκφραστεί επανειλημμένως και από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ιαπωνία. Έγινε μια συνάντηση της αποπτικής ομάδας χθες, όπου συζήτησαν με τον κύριο διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συζητήθηκαν λοιπόν οι διαπραγματεύσει που αποφασίστηκαν λίγε εβδομάδε εβδομάδες πριν. Η ο εισηγητής είναι ο Μέτιν Καζάκ. Σα ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντω, χθε έγινε αυτή η συνάντηση τη εποπτική ομάδα. Συζητήσαμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία για την ε, υπογραφή ενός ε, συμφωνού ελεύθερου εμπορίου. Συμμετείχαν οι συναδέλφοι από τη ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Εμπορίου και η συζήτηση ήταν άνοιχτη και αρκετά ενδιαφέρουσα. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στις 25 Μαρτίου φέτος. Θα γίνει μια ε, διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας και ο πρώτος ε, γύρος λοιπόν θα αρχίσει τον Απρίλιο. Έτσι αναμένεται. Ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης μας ενημέρωσαν ότι η αλλαγή της κυβέρνησης στην Ιαπωνία δεν θα έχει καμία επίπτωση στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει, παραμένει μια προτεραιότητα των ε, εξωτερικών σχέσεων της Ιαπωνίας. Επίσης, αναφέρθηκαν ορισμένα δασμολογικά εμπόδια και Υπόθηκε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην άρση των εμποδίων αυτών. Υπάρχουν βέβαια ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά εμείς χαιρετίζουμε την απόφαση της ε, Ιαπωνίας για την απαγόρευση εισαγωγών βοήου κρέατος, για την απόφαση άρσης λοιπόν της απαγόρευσης εισαγωγής βοήου κρέατος από τις κατοχώρες. Θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις που έχουμε ενώπιον μας δεν είναι εύκολες, σίγουρα είναι πολύπλοκες και υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι διαφωνίας πάνω σε πολύ σημαντικούς βασικούς τομείς στις εμπορικές μας σχέσεις. Για παράδειγμα, για τα ε, μη δασμολογικά εμπόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενδιαφέρον και έχει μεγάλες απαιτήσει όσον αφορά την παρασκευή τροφίμων. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις αιτήσεις ρήτρε. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν ορισμένε από αυτές. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε επαρκώς και δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτές. Πρώτα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ήμουν εκεί ως ε, σκιώδης εισηγητής της πολιτικής μου ομάδας. Να σας πω και εγώ λοιπόν ότι Εμείς καταδικάσαμε το, την πρακτική της ε, Ιαπωνίας για την ε, άρση. Εμείς μάλλον, όχι, εμείς ε, χαιρετίζουμε την ε, απόφαση λοιπόν της Ιαπωνίας για την άρση των δασμολογικών ε, εμποδίων και πιστεύουμε πως αυτό είναι ένα βήμα προς την γρήγορη ολοκλήρωση του ζητήματο αυτού. Έπειτα να πω ότι στο τέλος του προηγούμενου μήνα συναντηθήκαμε. Ο Φρανκ Προύστ ήταν εκεί, ο εισηγητής μας. Να σας ακούσουμε λοιπόν. Effectivement, c'était la première réunion constitutive de ce groupe entre l'Union européenne et Taïwan qui a eu lieu, qui a eu lieu donc le, le 30 janvier dernier. Euh, je voudrais simplement rappeler que nous avons souhaité euh,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 Uh, finally, Russia. Our monitoring, our standing rapporteur is Robert Sturdy, here on the table. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε επιτέλους η Ρωσία. Ο Τζόρτζ ήταν εκεί και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση και παρά το γεγονός ότι Έγινε μια πρώτη αδειολογία απόψεων ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν και ο αρμόδιος εκεί για την ε, Συμφωνία Εμπορίου με τη Ρωσία. Στη συνέχεια μίλησε ο κύριος Βλάντιμιρ Τσίζοφ και ρωτήσαμε τον κύριο Τσίζοφ αν μπορεί να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο δεν είχαμε ζητήσει αρχικώς. Έμεινε εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως αποδείχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ιδιαίτερε ανησυχίε για το τι ακριβώς ε, θέλει να κάνει η Ρωσία με τον ΠΟΕ. Ε, δεν θα τους εκπλήξει καθόλου να υπάρξει κάποια δράση κατά της Ρωσίας στο εγγύς μέλλον, παρά το γεγονός ότι δεν ε, επεκτάθηκαν περαιτέρω κυρίως συζητήσαμε πώς έχει κατάσταση για τις διαπραγματεύσεις και τα κεφάλαια της Νέας Συμφωνίας. Όπως γνωρίζετε, μόλις εντάχθηκε στον ε, ΠΟΕ η Ρωσία. Συζητήσαμε μία σειρά από ε, NTBs, ε, ε, τέλη ανακύκλωσης, άνθρακα, εξαγωγές, δυσανάλογα μέτρα φυτοϊγεία και κτηνιατρικά, SPS και φυσικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εισαγωγή στη Ρωσία ζών των ζώων σε καμία, από καμία χώρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή. Κατόπιν συζητήθηκε το θέμα των υπνοβηματοδών ποτών αλκοολούχα ποτά, διότι είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλη αγορά. Ο πρέσβης βέβαια δεν μπόρεσε να απαντήσει στην ερώτησή μου. Τον ρώτησα για τους ε, δασμούς εινοπνευματοδών ποτών ε, για την εισαγωγή στη Ρωσία. Ε, μου... Δεν μου απάντησε. Έκτοτε του απέστειλα επιστολή και μόλις μου απαντήσει επισήμως θα την διανύμω στην Επιτροπή για να την διαθέτετε και να διαβάσετε. Κάθε φορά, δύο φορές βέβαια συναντηθήκαμε, Κάθε φορά όμως λέει ότι τα μέλη της κάτω βουλής, της Δούμας, ε, είναι κατά της ε, αίτησης ε, της Ρωσίας για ένταξη στον ΠΟΕ και ορισμένες φορές χρειάζεται να δώσει μάχη με τους συναδέλφους στην κάτω βουλή που δεν θέλουν καμία σχέση με τον ΠΟΕ. Η επόμενη συνεδρία είναι για το Μάρτιο. Έχουμε προσκαλέσει τον κλάδο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσώπους τους για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και ο κύριο Τσίφ είπε ότι μία από τι βασικέ εξαγωγέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ρωσία είναι η ενέργεια. Ε, σχόλια από πλευρά σα, κύριε Πρόεδρε. Σχόλια, ερωτήσει. Ο κύριος Κουτάς. Ε, μία σύντομη παρέμβαση για να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Στάρντι πρέπει να πω ότι εξέπληξε ακόμα και μένα το γεγονός ότι ο πρέσβης είπε ότι το βασικό πρόβλημα σε αυτή τη στιγμή είναι και παραθέτω το πώς θα χωνέψουμε εντό εισαγωγικών την ένταξή μας στον ΠΟΕ και το ρωτήσαμε τι εννοεί με αυτή την έκφραση και μας εξήγησε τι έχει να πει και πρέπει να πω ότι μας ανησυχεί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία Ελπίζουμε όμως ότι εν τέλει θα καταλήξουμε στους απαραίτητους συμβιβασμούς για να προχωρήσουμε. Είμαι πολύ επιφυλακτικός όμως, δεν ξέρω κατά πόσον θα συμβεί. Είναι πολύ καλή πρωτοβουλία για την επόμενη συνεδρίαση, να γίνει μια συνεδρίαση και με την Gazprom. Ο Ρόμπερτ ε, κάνει καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Ρωσία τον Οκτώβριο και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά που θα έπρεπε να μας ανησυχούν για τη Ρωσία και ευχαριστώ ιδιαίτερα την ομάδα παρακολούθησης που παρακολουθεί τι συμβαίνει και ίσως αργότερα να μπορούσαμε ίσως να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή για να δούμε τι δυσκολίες ε, αντιμετωπίζουμε με τη Ρωσία. είναι πολύ σημαντικές ε, και πρέπει να τις συζητήσουμε. Στη συνέχεια έχουμε την Ινδία. Η Μαρία Μπαντία όμως, ε, η οποία είναι η μόνιμη συγγήτρια, δεν μπόρεσε να είναι παρούσα. Τη συνάντησα σήμερα το πρωί και αναχωρούσε για τη Βαρκελόνη, γιατί πρέπει να κάνει κάποια μικρή επέμβαση και ζητά συγγνώμη. Θα ε, είναι εδώ στην επόμενη συνεδρίαση και θα μας πει για τις τελευταίες εξελίξεις με την Ινδία. Θα πρέπει βέβαια να ακούσουμε τι έχει να μας πει, διότι η συνεδρίαση ήταν με τον κύριο Γκαρθία, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις με την Ινδία και όπως γνωρίζετε είναι βάσιμες οι ανησυχίες μας για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την Ινδία και νομίζω ότι θα πρέπει ε, να επανέλθουμε στην συνεδρίαση της ε, ομάδας παρακολούθησης με την Ινδία στην επόμενη συνεδρίαση. Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όχι. Ωραία. Να πω δύο πράγματα εγώ. Οι ομάδες παρακολούθησης, κατά την άποψή μου, είναι μια πολύ επιτυχής πρωτοβουλία της Επιτροπής μας. Θα ήταν αδύνατον ε, η Επιτροπή να παρακολουθεί αυτό που κάνουν οι ομάδες παρακολούθησης. Ε, συγκεντρώνουν πληροφορίες, εμπειρογνωμοσύνη και πρωτίστως ε, είναι ε, σε επαγρύπνηση για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει και παρακολουθούν στενά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο όφελος αυτών των ομάδων. Ε, δεύτερον, εργάζονται πάρα πολύ καλά κατά κανόνα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μόνιμους συζητητές. Επίσης, ε, να πω ότι θα ήθελα και οι σκιώδεις συζητητές ε, να ε, συμμετέχουν πιο ενεργά στις συνεδριάσεις. Βεβαίως και είναι εκεί η βοηθή τους και οι πολιτικοί σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων είναι παρόντες. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά όταν ε, έχουμε σημαντικούς προσκεκλημένους όπως ε, τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ανθρώπους από εξωτερικούς φορείς, ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και μια προσπάθεια να είναι παρόντες και σκιώδεις εισηγητές. Και μόνο για σεβασμό προς ε, τους προσκεκλημένους μας όσο σημαντικός και να είναι ο ρόλος ε, των μόνιμων εισηγητών, ο ρόλος των σχεδόν εισηγητών είναι εξίσου σημαντικός. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και είμαστε και εν αναμονή των εκθέσεων των υπολείπων ε, ε, ομάδων παρακολούθησης στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ε, όσοι λοιπόν δεν πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα για τη συνεδρίαση των δονηστών, παρακαλώ να αποχωρήσουν. Και επειδή έχουμε και 10 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών και θα ήθελα οι συντονιστές των ομάδων να ετοιμαστούν εντωμεταξύ για να ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών.